Θα ήθελα παρακαλώ να ζητούσω τους τέος πρόεδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κάτσουν εδώ στις ε, πολυθρόνες κάτω. Τους τέος προέδρους και τι τέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, ελάτε και καθίστε εδώ μπροστά. Και για εσάς υπάρχει μια ειδική έδρα εδώ, κύριε Πρόεδρε Πέτεριν Κόξ, κυρία Φοντέιν. We would like to start together with you. Να αρχίσουμε μαζί σας. we are hosting seven 7 πρώην προέδρους. Ο κύριος Μπορέλ έρχεται. Σας καλωσορίζουμε όλους. Okay, President Hans. κύριος Χένς. President Pat Cox. Ο κύριος Pat Cox. ο πρόεδρος Pat Cox. Okay. In a couple okay. of minutes they will be here. Two, three minutes. And... but... Δύο-τρία λεπτάκια και η κυρία Φοντέιν θα είναι εδώ και θα είναι μαζί μας και ο Ενρίκη Μπαρόν Κρέσπο. Έρχονται, είναι καθοδόν. presidents. Δεν θα γίνει δεύτερος γύρος ε, ψηφοφορίας, επομένως ε, έχουμε το χρόνο να περιμένουμε λίγα λεπτά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πέραν του γεγονότο ότι δεν περιμένουμε για να διεξαχθεί ο δεύτερος γύρος ψηφοφορίας. Δύο λεπτάκια λοιπόν δεν έχουν και τόση σημασία αγαπητοί φίλοι. Η κυρία Πρόεδρος Φοντέιν και ο κύριος Ενρίκε Μπαρόν Κρέσπο, πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Δύο πρώην Πρόεδροι, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ο οίκος σας, άλλωστε. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσει η συνεδρίασή μας μετά την διακοπή. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων 699. Λευκά και άκυρα 29. 670 λοιπόν έγκυρα. Η απόλυτα πλειοψηφία είναι 330. 336. 336 ψήφοι. Ο κύριος Ντεβά πήρε 142 ψήφους. Pan, pan Martin ο κύριος Μάρτιν Σούλτς. 387 ψήφοι. Η κυρία Νταϊάννα Ούολης. 141 ψήφους. Pan Martin... Ο κύριος Μάρτιν Σούλτς πέτυχε την απόλυτη πλειοψηφία των γύρων ψηφοδελτίων. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Congratulations. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια Πρόεδρε κύριε Σούλτς. Είμαι σίγουρος από τη δική σας ηγεσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα παραμένει το, ο κεντρικός παράγοντας της ε, ε, Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Εμείς ως βουλευτές έχουμε την υποχρέωση οι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν σε αυτά που κάνουμε. Όλοι εμείς υπολογίζουμε σε εσά κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει ως έχει στην καρδιά των συζητήσεων στην Ευρώπη και εκεί που γίνεται πολιτική προ όφελο των πολιτών της Ευρώπης. Θα ήθελα να σας καλέσω τώρα κύριε Πρόεδρε Σούλτσε να έρθετε στο Προεδρείο και να με αντικαταστήσετε στην έδρα ως νεοεκλεγής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.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 Αξιόλογες κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ για αυτό το αδιαφεσβήτητο αποτέλεσμα. Για τους περισσότερους από εσά μέχρι τις εκλογές αυτές ήμουνα πρόεδρος μιας άλλης πολιτικής ομάδας. Μιας πολιτικής ομάδας εδώ στο σώμα. μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείξατε σήμερα με τιμά. Θα εργαστώ πάθη θεία να μην απογοητεύσω την εμπιστοσύνη σας και να δώσω ισχυρή φωνή στο κοινοβούλιο μας. Θέλω το αξίωμά μου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να το ασκήσω έτσι, ώστε εκείνοι που με εξέλεξαν να μπορούν να είναι περήφανοι για την εκλογή που έκαναν και εκείνοι που δεν εξέλεξαν να είναι θετικά εκπλαγμένοι. Θα προσπαθήσω να είμαι ο πρόεδρος όλων των βουλευτών και θα προασπίζω κυρίες και κύριοι τα δικαιώματά σας. Καταρχήν όμω, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εσά, Πρόεδρε κύριε Μπουζέκ. Ήσασταν ο, πρόεδρο, ο πρώτος πρόεδρος του Θεσμικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίο προέρχεται από τα κινήματα υπέρ τη ελευθερία τη Ανατολική Ευρώπη. Και με την εκλογή σα και με τον τρόπο με τον ασκήσατε το αξίωμά σα, αποδείξατε τη νίκη της δημοκρατίας, τον θρίαβο της δημοκρατίας επί της δικτατορίας με την αξιοπρέπεια να χρησιμοποιήσατε το σώμα, προωθήσατε και αποδείξατε την ενότητα της Ευρώπης όπως κανείς άλλος πριν από εσάς. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναλαμβάνω το αξίωμα αυτό με μετροφροσύνη σήμερα. Η Ευρώπη διέχεται μια θελώδη περίοδο. Για πολλούς η καιρή είναι δύσκολη. Οι γονεί μου ανήκαν σε μια γενιά ακόμα που πίστευε ότι θα πρέπει τα παιδιά μας να ζούσουν καλύτερα από ότι εμείς. Και εμείς ζούμε καλύτερα. Όμως δεν έχουμε πια την βεβαιότητα ότι τα δικά μας τα παιδιά θα ζήσουν τόσο καλά κάποια στιγμή όπως εμείς. Οι επιπτώσεις της ε, οικονομικής κρίσης οδήγησαν σε αύξηση της φτώχειας σε πολλές χώρες και η ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων, έχει φτάσει σε δραματικά επίπεδα. Οι νέοι διαδηλώνουν στους δρόμους Ευρώπης κατά ενός οικονομικού συστήματος στο οποίο ορισμένοι λίγοι έχουν το κέρδος και οι απώλειες τις επομίζονται όλοι. Ακριβώς είδαμε τους τελευταίους μέρες ε, ανώνυμος οίκος αξιολόγηση Νέα Υόρκη να είναι πιο ισχυρή από ότι δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια και κυβερνήσεις. Θα πρέπει να τους ανητάξουμε ένα έντονο όχι. Γιατί αυτό οδηγεί σε μια κρίση εμπιστοσύνη στους θεσμούς της ε, Ένωσης. Ε, κρίση εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Αυτή η κρίση εμπιστοσύνη απειλεί, το πιστεύω, σε ε, το σχέδιο αυτό της Ευρώπης. Πολλοί παρακολουθούν το έργο μας με καχυποψία. Δεν ξέρουν αυτά που κάνουμε εμεί είναι σωστά. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι πολίτε της Ευρώπης δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για θεσμικέ συζητήσει, Ανησυχούν κυρίω για τη θέση εργασία του, για τη σύνταξή του, για την κοινωνική δικαιοσύνη, Θέλουν υγιή τρόφιμα, ε, καθαρό περιβάλλον. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε προσεκτικά να ακούμε τους ανθρώπους αυτούς. Καλύτερα να τους ακούμε. Γιατί εδώ ακριβώς ε, βρισκόμαστε στη, στον τόπο στον οποίο εκπροσωπούνται οι πολίτες της Ευρώπης. Εμείς εδώ είμαστε οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού. Και γι' αυτό σας λέω, ότι προς τους πολίτες που μας έχουν σε άμεση ψηφοφορία εκφράσει την εμπιστοσύνη τους δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Περιμένουν από εμά να προσπίσουμε τα συμφέροντά τους. Με περηφάνεια μπορώ να πω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ στο ε, σώμα είναι οι συνήγοροι των εκλογέων τους και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους. Αλλά για πρώτη φορά κυρίες και κύριοι από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ληστικό σενάριο. Εδώ και μήνες η Ένωση κινείται από μια διάσκεψη κορυφής κρίσης στην άλλη. Αποφάσεις μας αφορούν όλους. Κάθε έναν από εμά εδώ στην αίθουσα, κάθε έναν πολίτη λαμβάνονται από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και κλεισμένων των θυρών. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι μια η σε εποχές που δεν τις ε, ε, θέλουμε να ξανάρθουν. Θυμίζει την εποχή του συνεδρίου της Βιέννης τον 19ο αιώνα. Τότε αξίωμα της πολιτικής ήταν σκληρή επιβολή των εθνικών συμφερόντων και χωρίς κανένα δημοκρατικό έλεγχο. Απ' την άλλη μεριά όμως η Ευρώπη της μεταπολεμικής εποχή στηρίζεται στη ρεαλιστική αντίληψη ότι οι συμφέροντά μα δεν μπορούν να διαχωριστούν από τα συμφέροντα των γειτόνων μα. Βασίζεται στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ένα παιχνίδι μηδενικού αστρίσματο το οποίο κάποιο πρέπει να χάσει για να κερδίσει κάποιο άλλο. Ακριβώ το αντίθετο. Ή όλοι θα χάσουμε ή όλοι θα κερδίσουμε. Ο βασικός κανόνας εδώ είναι η κοινωτική μέθοδος. Αυτό δεν είναι μια τεχνική έννοια. Η κοινωνική μέθοδος είναι η ψυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Σημαίνει ότι οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με διάλογο και συνένεση. Αντί να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου, να επικρατούν η ελληνική και η δημοκρατία. Να επιτευχθεί ισορροπία συμφερόντων μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών, μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολή και Δύση και ιδίως να προωθηθεί η ευημερία όλων και να τη βάλουμε αυτή πάνω από τα ατομικά συμφέροντα. Αυτό σημαίνει ε, κοινοτική μέθοδος. Αυτό κυρίες και κύριοι πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, ήταν αυτονόητο και επιτυχές εγχείρημα. Όμως, αυτό το κοινοτικό σχέδιο επλήγει. Τα δύο τελευταία χρόνια δεν άλλαξε μόνο ο τρόπος ε, ε το ίδρα των προβλημάτων, αλλά και η μέθοδος αντιμετώπισης τους. Γιατί η παραπομπή των θεμάτων συναντήσει κορφή και διαρκώ περισσότερη συναντήσει αρχικών κυβερνήσεων και αστείωση σε αυτέ αποκλείουν σε μεγάλο βαθμό από τι διαδικασίε λήψη αποφάσεων το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο τη κοινότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων υποβαθμίζουν ουσιαστικά σε εκτελεστέ αποφάσεων. Γιατί το μόνο που του απομένει είναι να συγκατανεύουν τι κυβερνητικέ συμφωνίε. Σα λέω όμω το αποτέλεσμα μια ανεπαρκώς βασισμένη στην κοινοβουλευτική άποψη πολιτικής θεωρείται από του πολίτε ω διαταγή από τι Βρυξέλλε. και αυτό το πληρώνουμε όλοι, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δημιουργείται έτσι ένα γόνιμο έδαφος για να πηχθούν αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα παρακολουθεί αυτή την κατάσταση άπραγο, ελπίζω. Μπορούμε να, να έχουμε περισσότερη Ευρώπη με λιγότερο κοινοβουλευισμό. Όχι. Αυτούς, αυτούς τους ανθρώπους που αυτό προσπίζουν θα τους μαχηθούμε και εγώ με σας όλοι μαζί. Η διακρατική συμφωνία για μια νέα δημοσιονομική ένωση αποτελεί μια πρώτη δοκιμή. Στι διαπραγματεύσει αυτέ, οι εκπρόσωποι του κοινοβουλίου μα, Φερχόφστατ, Μπροκ, Γουαλτιέρη και Κονβέντιτ, με την απέτησή τους, με την απέτηση του Κοινοβουλίου να υπάρχει λιτότητα δημοσιονομική αφενός και από την άλλη ανάπτυξη και απασχόληση, ήταν καταρχήν χωρίς αποτέλεσμα. Αλλά τώρα κάτι κινείται με την πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ελπίζω ότι αυτή η ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχία και ανάπτυξης είναι αυτό ακριβώς που θέλουν οι πολίτες. Και για να πετύχει αυτό θέλω στις ε, κορυφή κορυφής να είναι και το Κοινοβούλιο στο τραπέζι των πραγματεύσεων. Δεν μπορούν να καλούνται όλοι εκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρώπη, κυρίε και κύριοι, είναι μια κοινότητα αξιών. Από τι ψήφιε χώρε απαιτούμε την αυστηρή τήρηση των ε, κριτηριών τη Κοπενχάγη. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αγωνιστεί για να εξασφαλίσει και στα κράτη-μέλη να τηρούν και να εφαρμόζονται ω αυτονόητε αξίε η δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίε. Όποιο παραβιάζει τι αξίε του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξέρει ότι θα είμαστε έντονα αντίθετοι. Έχουμε την υποχρέωση αυτή αναλάβει ω Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προσθέσω κάτι πολύ επίκαιρο. Αύριο θα έχουμε μια πολύ ανηφατική συζήτηση για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ο Πρωθυπουργό Όρμπαν ε, ενημέρωσε τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι αύριο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα παρουσιάσει δική του άποψη της κατάστασης. Εγώ ήρθα στη διαβούλευση με τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων και θα διαβουλευτώ και με εκείνους που δεν μπορούσα ακόμα να διαβουλευτώ μαζί τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνουμε, να δεχθούμε την παράκληση αυτή του κυρίου Όρμπαν, αν συμφωνεί η Ιδανική Προεδρία, να του δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσει εδώ και να παρουσιάσει τη δική του άποψη. Γιατί ακριβώς αυτό εννοώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει αντιφατικές συζητήσεις για την κατάσταση στην Ευρώπη. Και γι' αυτό καλό θα είναι να έρθει ο κύριος Όρμπαν εδώ αύριο. Και μου φαίνεται ότι καλό ε, τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει η ε, Κομισιόν στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Πολιτών να συζητούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ακούμε και την αντιπολίτευση κοινωνικών πολιτών της ε, ε, Ουγγαρίας. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ε, είναι σωστό ένα επικεφαλή ενό κράτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν εδώ, σε εμά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το καθήκον του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ω Προέδρο ενό των και κεντρικών θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι είναι να ενταχθώ σε αυτή την συνεχιζόμενη τάση στις συνόδους κορυφής και στην επανεθνικοποίηση. Θέλω να συμβάλλω το Κοινοβούλιο να είναι πιο ορατό και να ακούγεται περισσότερο χώρος της δημοκρατίας και του πολυφωνικού διαλόγου. Πρέπει να δίνουμε στα λόγια μας, κυρίες και κύριοι, μεγαλύτερο βάρος. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να βρισκόμαστε επίση όρει με το Συμβούλιο στι διαπραγματεύσει του μαζί του. Είτε αυτέ αφορούν τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, είτε μεταρρύθμιση γεωργική, αλληλευτική ή περιφερειακή πολιτική, τον αγώνα κατά τη αλλαγή του κλίματο, την ε, θέσπιση νομοθεσία για τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, την δικαιοσύνη, τι εσωτερικέ υποθέσει ή την εμπορική πολιτική. Έχει τεράστια συμπληρωματική ευθύνη αναλάβει πια το Κοινοβούλιο. Εδώ και δύο έτη έχει τεθεί σε εφαρμογή συνθήκη Λισαβόνα που πιστεύω δεν έχουμε ακόμα α, εκμεταλλευτεί πλήρως εμείς ως πρώτου του λαού. Πρέπει να είναι κοινό μα στόχο η αξιοποίηση των πραγματικών μα αρμοδιοτήτων. Ακόμα και αν χρειαστεί να έρθουμε σε σύγκρουση για να το πετύχουμε. Για να ενισχυθεί η ορατότητα του έργου του Κοινοβουλίου, απαιτείται επίση κριτική εξέταση των συμφωνών πρώτη ανάγνωση. Χρειαζόμαστε συζήτηση και για τη δική μας εργασία. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν υπάρχει τάξη στο ίδιο το σώμα. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια με τη βοήθεια της διοίκησής μας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί τα κοινοβουλευτικά όργανα και όλοι οι βουλευτές να έχουν εκείνο το πλαίσιο στο σώμα που είναι απαραίτητο για την βέλτιστη εκτέλεση των καθηκόντων τους ως νομοθετών. Κυρίε και κύριοι, δεν θα είμαι εμβολικό πρόεδρος. Θα είμαι ο πρόεδρος που θα μαχηθεί, αν χρειάζεται, για να διασφαλίσει η εκτελεστική αξία να κερδίσει το σεβασμό του Κοινοβουλίου. Ένας πρόεδρος που ε, <clears throat> θα προσπίζει τα συμφέροντα των πολιτών. Ένας πρόεδρος που εκπροσωπεί ισχυρούς βουλευτέ που αγωνίζονται για τα συμφέροντα των εκλογέων του. Ένα πρόεδρος που θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ξανακεργηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών στην διαδικασία Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Και θα προσπαθήσω να αναζωπηρώσω τον ενθουσιασμό για την Ευρώπη. Σύντροφοι, πολλοί έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Πολλοί έδωσαν τη ζωή τους υπέρ των κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων και του κοινοβουλευτισμού. Ο πρώτος ελεύθερα εκλεγμένος προέδρου της συντακτικής συνέλευσης στην Ισία, ο Μουστάφα Μπεντζαφά, με τους συναδέλφους του, που βιώνουν την πρώτη κοινοβουλευτική εμπειρία έχουν στραμμένα τα μάτια τους προς τα κοινοβουλία στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην Λιβύη, όπως ένα, ένας ε, δυνάστης δεξίχα πόλεμο κατά του ίδιου του λαού του, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτη άνοιξε πρεσβεία και έδωσε έτσι ελπίδα στους ε, ανθρώπους που βρίσκονται εκεί σε τόσο δύσκολη κατάσταση. Όταν ε, απονημήθη το βραβείο Ζεχόροφ πριν από μερικέ μέρε, μια θαραλέα νεαρή blogger και ένα συλλογικό αντίπλο του Καντάφη μα συγκίνησαν με τον θαυμασμό που εξέφρασαν για τι εξή τη Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή μα ρωτούν επανειλημμένα πώ κατορθώσαμε στην Ευρώπη να μετατρέψουμε εχθρού σε φίλου. Και πώς μπορέσαμε πέρα από τις εθνικές και θρησκευτικές ε, διαφορές να οικοδομήσουμε αυτή την μία Ευρώπη. Όσο περισσότερο απομακρύνεται κανείς γεωγραφικά από την Ευρώπη, τόσο πιο ενθουσιασμό ε, ακούει για το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ας ξαναφέρουμε αυτόν τον ενθουσιασμό πάλι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια ιδέα συναρπαστική. Μια ιδέα που δημιουργήθηκε σαν απάντηση του δεύτερου ημισεως του 20ου αιώνα στο πρώτο ημισή του ίδιου αυτού αιώνα. Ποια μορφή είχε το πρώτο του 20ου αιώνα. Μίσος. Πολιτική μεγάλων δυνάμεων. Διώξεις κατά άλλων. Περιφρόνηση των ατόμων. Χαρακόπητο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Τα γκούλακ του Στάλιν. Και Θαλαμεριού του Άουσβιτς. Οι πιο μαύρες ιστορίες, ε, σελίδες συγγνώμη, της ιστορίας του πολιτισμού. Στο δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και τα κοινά θεσμικά όργανα της Ευρώπης της εξασφάλισαν τη μακρύτερη περίοδο ευημερίας και ειρήνης της ιστορίας της. Το 1989 έπεσε το Σιδηρούν παραπέτασμα. Επανώθηκε η Γερμανία. Το 2004 και το 2007 προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώην κράτη του Συμφώνου της Βαρσοβίας και με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε και πάλι πολιτιστική και πολιτική ενότητα της Υπήρου που ήταν τεχνητά χωρισμένη επί 40 χρόνια. Πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό. Γιατί πάσαμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Γιατί επιτρέπουμε να ακούγονται αρνητικά σχόλια για το μοναδικό αυτό ιστορικό επίτευγμα. Κυρίες και κύριοι, ο παππούς μου αγωνίστηκε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 20 χρόνια μετά ο πατέρας μου ε, πήγε σε ένα πόλεμο, άλλο σε ένα πόλεμο με το οποίο ο Χίτλερ έκαψε όλο τον κόσμο. Εγώ μεγάλωσα σε μια μικρή χώρα στα σύνορα που οι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν ώρες στα σύνορα για να πάνε να επισκεφτούν τους φίλους τους στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία. Ξεπεράσαμε τον πόλεμο και την πείνα, ανοίξαμε τα σύνορα, καταδικάσαμε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ζούμε σήμερα σε μια ελεύθερη, σε μια ανοιχτή Ευρώπη. Μια Ευρώπη που μπορεί να είναι περήφανη για την πολιτιστική της πολυμορφία. Ας οπλίσουμε αυτή την Ευρώπη για τον 21ο αιώνα, ούτω ώστε και η νέα γενιά, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών, να δούνε στην Ευρώπη αυτή μια υπόσχεση για οικονομικά δυνατή κοινωνικά δίκαιη, ελεύθερη και δημοκρατική ευρωπαϊκή πατρίδα. Αυτό είναι το κοινό μας έργο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.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 Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω. Η ημερησία αναδιάταξη προβλέπει τώρα. Προβλέπει ένα γύρο των προέδρων των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα καταρχήν να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Ιωζεφ Τόλεξ, ονόματο του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητέ Μάρτιν, αγαπητοί συνάδελφοι, εξ ονόματος του ΕΛΚ και προσωπικά. Θα ήθελα να σε συγχαρώ και να συγχαρώ τον νέο μας πρόεδρο. Του εύχομαι. Κουράγιο. Διάβια πνεύματος και δύναμη ώστε να μπορέσει το όργανο το οποίο εκπροσωπεί συλλογικά 500 εκατομμύρια πολίτες να συνεχίσει να εργάζεται με τον τρόπο που εργάζεται. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τον Μύρ Σουντεβά και την Διάννα Βόλις που ήταν επίσης υποψήφοι για την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να του πω ότι παρά το γεγονό ότι τα δύο μεγάλε πολιτικέ ομάδε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή τη θητεία είχαν αποφασίσει να ασκήσουν την Προεδρία διαδοχικά αυτή την θητεία, θα ήθελα και εγώ να του συγχαρώ διότι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία της εκλογής. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω σήμερα το πρωί Μάρτιν Σούλτς όλους τους Πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο Μπούζεκ που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, να επωφεληθεί από τις εξαιρετικές ικανότητες που είχε ως εργός κράτους, που είχαν επωφεληθεί οι Πολωνοί. Τον ε, πρόεδρο Πέτερν όλους τους ε, σα, σχίζοντα από την πρώτη πρόεδρο εξελέγει με καθολική άμεση ψηφοφορία την Σιμών Βέιλ. Όλου τους πρόεδρους οι οποίοι διαδέχτηκαν ένα άλλο εδώ και ενίσχυσαν τι αρμοδιότητε και την ε, όλη εξουσία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε Σούλτ, και εσεί θα συνεχίσετε. Τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε ω Πρόεδροι πολιτικών ομάδων να συνεργαστούμε. Οι πολιτικέ σα πεπιθήσεις περισσότερες οποίε δεν συμμερίζονται και οι πολιτικές μας ομάδες αποκλίνουν σε πολλά θέματα. Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να σας έχουμε εμπιστοσύνη, διότι σε δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει σήμερα την Ευρώπη, αυτό το οποίο μας ενώνει είναι πολύ περισσότερο σημαντικό από αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι είσαστε αποφασισμένος να προασπίσετε τα γενικά συμφέροντα της Ευρώπης Μπροστά στην πολυμορφία των εθνικών συμφερόντων, η πολιτική μου ομάδα δεν μπορεί να σα υποστηρίξει πλήρω σε αυτή την δράση, σε αυτή την αποστολή, έχοντα συνείδηση ότι οι επόμενοι μήνε θα είναι μία από τι πιο ε, κρίσιμε περιόδου που γνώρισα από τη δημιουργία τη Ευρώπη. Έχετε, κατά την άποψή μα τρει προτεραιότητε. Την κοινοτική μέθοδο να την προασπίσετε, να την ε, ε, υπερασπιστείτε και να την διασφαλίσετε. Επίσης, θα πρέπει το γενικό συμφέρον της Ευρώπης να το προσπίσετε, να μπορέσετε να, προσ... να προστατεύσετε τις μικρές, τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης και να μην ε, επιτρέψετε σε κανέναν να μείνει ε, χωρίς να ενεργεί στη θέση του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενεργούμε ενισχυμένοι στην Ευρώπη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Τίποτα είναι πιο σημαντικό που να αποδείξουμε στους πολίτες μας ότι το ευρώ θα είναι ένα ισχυρό νόμισμα που θα διαρκέσει. Αυτό εάν κάνουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε από την ε, δημιουργία του. Δηλαδή να έχουμε και πολιτική και οικονομική διακυβέρνηση. Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από το να διασφαλίσουμε το κοινό αγαθό που είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των 550 εκατομμυρίων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, δημιουργώντας αυτό το οποίο θα έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πατέρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν μία πρωτοβουλία όγνωρη κρίση, δηλαδή καθόρισαν την ε, μοίρα των ε, λαών, ενώνοντας τους λαοί οι οποίοι ε, αλληλοσκοτώνοντας το παρελθόν. Ο Ντεγκάσπρο, ο Ντανάουερ και όλοι οι παιδές της Ευρώπης σήμερα συνέχισαν το όνειρο της Ευρώπης παρά τις οικονομικές δυσκολίες και παρά το γεγονός ότι έχουν αλλάξει σε γεωστρατηγικό επίπεδο πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Είναι δικό μας καθήκον να μην τους απογοητεύσουμε, να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την πολιτική που κάνουμε για να ξεπεραστεί η κρίση και να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας όχι μόνο ένα βιώσιμο μέλλον, αλλά κυρίως ένα καλύτερο μέλλον. Εσείς κύριε Πρόεδρε λοιπόν και εμείς όλοι αγαπητοί συνάδελφοι ως εκπρόσωποι εκλεγμένοι των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά πρώτον αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Και εσείς και εμείς θα πρέπει να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με αίσθημα ευθύνης. Αποκινούμε την Κομισιόν που είναι η θεματοφύλαξη των συνθήκων, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σύγκληση οικονομική πολιτική. Αυτά είναι τα καλύτερα όπλα τα οποία θα έχουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση που διερχόμαστε. Αγαπητέ Μαρτίν Σούρπ, ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ανταποκριθεί σε πολλέ εξωτερικέ προκλήσει και το ΕΛΚ θα είναι πάντα μαζί σου για να μπορέσει σε πνεύμα ευρωπαϊκό να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει. Σε ενθαρρύνουμε επίση να μπορέσει αυτό το μήνυμα να το αποστείλει σε χώρε ε, όπως η Ουκρανία, όπου η Γιούλα Τιμουσέγκο αντιμετωπίζεται με παράδεικτο τρόπο, ή σε χώρες όπως η σε χώρε όπου η βούληση αλλαγής ε, ε, των πολιτών καταστέλλεται με παράδειγμα τρόπο. Επίσης, χαιρετίζω την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλεις για να αλλάξουν κάποια εσωτερικά πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα πρέπει ο κώδικας συμπεριφοράς να αλλάξει ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθύνη εκ μέλου όλων των κρατών των ε, μελών. Η, το, η πολιτική μου ομάδα σε υποστηρίζει. Αγαπητέ Πρόεδρε, εφ' εξή ηγείσαι ε, νου θεσμικού οργάνου που είναι μοναδικό στον κόσμο. Για δυόμιση χρόνια είσαι ο ηγέτη μια κοινοβουλευτική συνέλευση που δεν θέλει να επιβάλλει τίποτα αλλά να πείσει το Συμβούλιο ότι δημιουργώντα μια συνθήκη 2, μια διακυβέρνηση δύο και ένα κοινοβούλιο δύο θα αντιμετωπίσουμε τι παρούσες δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, σύσσωμοι μαζί σα, κάθε φορά που θα υπερασπίζεστε αυτή την ενοποιημένη Ευρώπη, αυτή την αλληλέγγυη Ευρώπη για να μπορέσουν να ευρεθούν καινοτόμε λύσει, θα είμαστε μαζί σου. Κάθε φορά που θα προασπίζεσαι τις κοινέ πολιτικές της Ευρώπης. Κάθε φορά που θα αγωνίζεσαι ώστε να υπάρχουν κατάλληλα κονδύλια για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές. Κάθε φορά που πέραν των συνόρων μας θα προασπίσει και θα προωθείς τα ιδεώδη και τις αξίες που διέπουν την ένωσή μας. Ανεκτικότητα, αλληλεγγύη και ελευθερία για όλους. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο εγχείρημά σου, αγαπητές πρόεδρε Σούλτς. Euh, Ευχαριστώ, συνάδελφε Ντόλ. Το λόγο έχει η από το Δημοκρατική Ομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος ε, της ομάδας των ε, προοδευτικών και σοσιαλιστών θα ήθελα να σε συγχαρώ με ιδιαίτερη θέρμη για αυτή την εκλογή σου ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σου πω ότι για την ομάδα μας είναι τιμή ένα αξιότιμο μέλος όπως εσύ να μας οδηγήσει σε αυτό το επόμενο βήμα εδώ στο Κοινοβούλιο σε μια στιγμή που το είπες και εσύ ε, που βιώνουμε πολλά προβλήματα, έχουμε πολλές απειλές και πολλούς κινδύνους και για την ίδια την Ευρώπη αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προβλήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανεργίας, ε, η οικονομική και η κοινωνική κρίση και επίσης ο κίνδυνος να χάσει τη βαρύτητά του το Κοινοβούλιο ε, λόγω αυτής της ε, κυβερνητικής στάσης, φονταμενταλιστικής στάσης. Και αυτό που βιώνουμε πιο ε, πολύ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή είναι η ανάγκη να έχουμε ειδικού ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν μεγάλη ευρωπαϊστική ε, δυνατότητα, ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μάχη και έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν ενός προγράμματος και αντίστοιχο πάθο. Και εσύ, αγαπητέ Πρόεδρε, είσαι ο άνθρωπο ο οποίο διαθέτει όλες αυτές τις ικανότητες. Ε, μπόρεσα να συνεργαστώ μαζί σου εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα και ξέρω γιατί ακριβώ μιλάω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινά αυτή η Προεδρία εντό όλων αυτών των συγκρούσεων, ώστε να μπορέσουμε με την ηγετικό σου ρόλο να δημιουργήσουμε μια νέα τάση για αυτή την Ευρώπη που χάνει λίγο το βηματισμό της. Ε, σήμερα δεν είσαι ο πρόεδρος της πολιτικής μας ομάδας, είσαι ο πρόεδρος όλων των εκπροσώπων εδώ του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα να σου επενθυμίσω τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό που προσπαθούμε και πάντα θα προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική, πιο ε, καλή Ευρώπη για όλους. Και να σου πω ότι γι' αυτό το στόχο θα μας βρεις πάντα δίπλα σου. Καλή τύχη και καλή τύχη στις εργασίες σου. Ευχαριστώ, συνάδελφε Μπαδιά. Το λόγο έχει εξ νόμου τη των Φιλελευθέρων, ο συνάδελφο Φεφόφστατ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Μάρτιν, εξ ονόματος της ομάδας μου και εξ ονόματος ε, δικού μου φυσικά συγχαρητήρια για την εκλογή σου, συγχαρητήρια και σε όλα ε, στους υπόλοιπους υποψηφίους ε, για αυτές τις εκλογές για τον Πρόεδρο και να πω ότι ε, απόλαυσα την πρώτη σας ομιλία κύριε Πρόεδρε. Ξεκινήσατε με λίγο σοσιαλδημοκρατικό τόνο αλλά στο τέλος πραγματικά μιλούσε ο ίδιος ο Πρόεδρος. Μαθαίνετε πολύ γρήγορα λοιπόν κύριε Πρόεδρε τα νέα σας καθήκοντα. Καταρχάς, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ε, μιλήσω στον προκάτοχό σας, τον κύριο Μπούζεκ, με τον οποίο συνεργάστηκα εδώ και αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μπορούμε να είμαστε μάρτυρες του γεγονότος ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι ήταν το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κάνατε αξιοσημείωτο έργο εδώ στο Κοινοβούλιο. Καταφέρατε να προσαρμοστούμε σε αυτή τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, που έπρεπε να εφαρμοστεί και ε, προσπαθήσατε μαζί με το Κοινοβούλιο να κάνετε όλες αυτές τις πολιτικές για την καταπολέμηση της κρίσης και εγώ χαίρομαι μαζί με τους υπόλοιπους Προέδρους τη διάσκεψη των Προέδρων που είχα τη χαρά να συνεργαστώ ε, μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για τα όλα όσα κάνατε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ότι στη διάρκεια της ε, εκστρατεία σα για την ε, Προεδρία του Κοινοβουλίου, άκουσα πολλού συναδέλφου που να λένε ότι ναι, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ουδέτερο πρόεδρο. Χρειαζόμαστε ένα πρόεδρο ο οποίο δεν θα ψηφίζει. Ένα πρόεδρο ο οποίος δεν θα έχει άποψη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ξεπλάγει από αυτές τις δηλώσεις. Εγώ είμαι της άποψης ότι χρειαζόμαστε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει άποψη και δεν είναι ουδέτερος, διότι δεν είναι δυνατόν τη σήμερα ημέρα κύριε Πρόεδρε να παραμείνουμε ουδέτεροι ε, ενώπιον ε, του φανταμενταλισμού που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Είναι αδύνατον, αγαπητοί συνάδελφοι, να μείνουμε ουδέτεροι ενώπιον ενός Συμβουλίου το οποίο κάθε φορά προσπαθεί να ε, υπονομεύσει την κοινοτική μέθοδο και τη μέθοδο την οποία ε, σκέφτηκε ο Ζαμονέ. Είναι πολύ δύσκολο να μείνουμε ουδέτεροι όταν κάποιο επιτίθεται στην κοινοτική μέθοδο και να γίνεται καθημερινά αυτό στο Συμβούλιο αλλά και εκτό Συμβουλίου. Και είναι αδύνατον να παραμείνει κάποιος ουδέτερος ενώπιον του εθνικισμού και του λαϊκισμού ο οποίος αυξάνεται στην Ευρώπη και δεν ανήκει στις ευρωπαϊκές μας αξίες. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να είστε ένας πρόεδρος, αλλά δεν θα ήθελα να είστε ένας ουδέτερος πρόεδρος. Χωρίς φίλο, ο οποίος δεν έχει άποψη. Το αντίθετο, εγώ θα ήθελα ένα πρόεδρο, αγαπητέ Μάρτιν, ο οποίος θα εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα εκπροσωπεί σε κάθε περίπτωση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα τα οποία διαφέρουν από τα συμφέροντα των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Θα ήθελα ένα πρόεδρο ο οποίο θα δώσει μάχη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και γιατί όχι να το πούμε χρειάζομαι ένα πρόεδρος ο οποίος θα είναι υπέρ της Ομοσπονδιακής Ευρώπης, της Φεδεραλιστικής Ευρώπης που επιθυμούσαν ο Μονέ, ο Σουμάν, ο Ντεγκάσπαρη και ο Σπινέλη. Και επιπλέον ή δυνατόν, αγαπητέ Μάρτιν, θα ήθελα ένα πρόεδρος ο οποίος θα εξηγεί στα κράτη-μέλη όταν πηγαίνει επί τόπου, διότι θα σε προσκαλέσουν ε, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με, ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δράξει τη δυνατότητα, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί σου, να πεις την αλήθεια στα κράτη-μέλη και να του πει ότι Πρόκειται για μια δημοσιονομική, οικονομική και πολιτική ένωση. Αυτή είναι η ένωση που θα μπορέσει να διασώσει το ευρώ. Και τέλος, η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει το δρόμο. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να αποδείξει ποιος είναι ο δρόμος για την κρίση. Και είναι απλό. Η Ευρώπη δεν είναι το πρόβλημα σε αυτή την κρίση. Η Ευρώπη αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα που ε, αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και τέλος, να δεχτείτε τους πρώην συναδέλφους, ε, ο επικεφαλής των ομάδων που ορισμένες φορές είπαν και κάποια κουβέντα παραπάνω, ε, νερό ναι, στο κρασί σας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Φαρουφστάτ. Εξ ονόματο τη ομάδα των Πρασίνων, η συνάδελφο Άρμ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Μάρτιν Σούλτ. Πρωτού περάσω στην... στα συγχαρητήρια, θα ήθελα καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω του προκάτοχου σου, ε, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που γνώρισα, όπω ο Γιάννη Μπούχο, ότι και ο Χάντ Κιάτ Πέτερινγκ και ο Σβερέλ πάντα είχαν τη δική τους μορφή για να αντιμετωπίσουν τις ε, ε, καθημερινές προκλήσεις. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και τους ε, άλλους υποψήφιους γιατί η εσωτερική δημοκρατία ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι. Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία είναι εκείνη που πέτυχες εσύ σήμερα και αυτό έχει τους λόγους του. Δεν ε, είναι επικεφαλής του σώματος σήμερα ένας σοσιαλδημοκράτης. Όχι, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας σοσιαλδημοκράτης ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός κοινοβουλευτικός. Ε, θα ήθελα να σου θυμίσω όταν ε, με ρώτησες τι θα πίστευα να γι... αν γινώσουν πρόεδρος του κοινοβουλίου ρώτησα Πώς ήρθε αυτό. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ τον Μάρτιν Σούλ σαν πρώτο εκπρόσωπο εδώ ε, και διπλωματικά περιορισμένο επικεφαλής του σώματος. Ενώ μεταξύ όμως το φαντάζομαι αυτό πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ελπίδα ότι την δική σου η ιδιαίτερη προσωπικότητα θα τη διατηρήσεις. Και η διπλωματική μορφή που καμιά φορά χρειάζεται διπλωματική συμπεριφορά δεν θα σε παρασύρει αλλά θα εξακολουθείς να είσαι ανοιχτός όπως γνωρίσαμε εδώ δύσκολος όπως γνωρίσαμε εδώ και στο νέο σου αξίωμα και αυτή την δύσκολη προσωπικότητα να τη χρησιμοποιήσεις και σε ε, αντιπαραθέσεις με τον κύριο Πρόεδρο Μπαρόζο αλλά και με τον Φανράμποϊ, με την ε, κυρία Μέρκε και τον κύριο Σαρκοζή. Η υπόσχεση που έδωσε στην προσωπική σου εκστρατεία ήταν καμιά φορά πολύ συγκινητικά απλοϊκή. Όλοι για τον έναν και αν λειτουργεί αυτό θα λειτουργεί και το ένας για όλους. Αυτή την προπόθεση δημιούργησε όμω σήμερα το Κοινοβούλιο. Τώρα έχουμε αντιπαραθέσει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να δούμε ότι δεν είναι μόνο ο νέος πρόεδρος του Κοινοβουλίου εκείνος που θέλει να ακολουθήσει μια νέα οδό στις αντιπαραθέσεις αυτές, αλλά και ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο είναι σε θέση να προωθήσει αυτούς τους στόχους που έχει μόνο του ορίσει. Ένα παράδειγμα μπορώ να σκεφτώ εδώ είναι η αντιπαράθεση με τον Βικτόρα Ορμπάν όπου η συζήτηση για, για την νομοθεσία για τα ΜΜΕ απέτυχε σε μια χρονική στιγμή στην οποία πολλά θα μπορούσαμε να πετύχουμε γιατί η τελευταία αναλύση το Κοινοβούλιο άφησε το θέμα στην Κομισιόν για να οργανώσει διαφορετικά την κατάσταση και να εξαφανιστούν τα προβλήματα. Αυτό δεν επιτρέπεται να ξαναγίνει στην περίπτωση της Ουγγαρίας και επειδή αναφέρθηκε και το όνομα της Βούλια Τιμοσέγκο που χειροκρότησα εγώ δεν επιτρέπεται σε ένα κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή κατά την οποία στην Ρωσία οι πολίτες εξακολουθούν ε, προσπαθούν συγγνώμη, να κινηθούν κατά της κατευθυνόμενης ε, δημοκρατίας σε μια περίοδο στην οποία οι Ουκρανοί είναι απελπισμένοι, δεν επιτρέπεται λοιπόν να αφήσουμε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωση να κινηθεί εκτός δημοκρατίας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή πάση θυσία και με τη βοήθεια του Πρόεδρου. Μάρτιν Σούλτς, αναλαμβάνει το αξίωμα αυτό κατά τη γνώμη μου, σε μια στιγμή η οποία είναι ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι είχε φανταστεί ότι θα ήταν πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι η τελευταία διάσκεψη κορυφής για την κρίση δεν θα είχε καμία επίδραση στις περαιτέρω εξελίξεις. Έρχομαι τώρα μόλις από την Ιαπωνία και είδα το γεν, το νόμισμα μιας χώρας με τεράστια προβλήματα, πώς το γεν λέω ανέ, ανέβηκε σαν κομίτης ξεπετάθηκε στα ύψη. Αυτό δεν είναι λογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν πρέπει να κατηγορούμε τους ε, οργανισμούς ε, αξιολόγησης, αλλά το ότι η πολιτική δεν έχει αρκετή επίδραση και ότι περισσότερη επίδραση έχουν αυτοί των μεγαλοτραπεζών, αυτές, αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης, είναι απαράδεκτο. δεν θέλω να πω ότι το Κοινοβούλιο αποτελείται πια από σοσιαλδημοκράτες, αλλά πολλέ από που ανέπτυξε το σώμα αυτό κατά της κρίσης με πλειοψηφία θα πρέπει να προωθηθούν έναντι του Συμβουλίου και της Κομισιόν μέχρι το τέλος. Δεν επιτρέπεται πριν ακουστούν οι ιδέες μας να ε, τις ε, ε, εγκαταλείπουμε και να προχωρούμε στον ε, επόμενο συμβασμό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία Μάρτιν ξέρω ότι θα είσαι δύσκολο. Για τη δική μου πολιτική ομάδα έχω να πω ότι και εμεί θα είμαστε μια δύσκολη πολιτική ομάδα. Και εξ ονόματο των γυναικών του σώματος εδώ θα ήθελα εδώ να πω ότι μετά την Σίμον Βέιλ και μετά την κυρία Φοντέν θα ήταν πολύ καλό εάν από σήμερα προετοιμάζαμε οι γυναίκες του Κοινοβουλίου ο επόμενος πρόεδρος στην επόμενη θητεία να είναι μία πρόεδρος γυναίκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Χάρμς. Το λόγο στον των συντηρητικών έχει ο συνάδελφος Κέλεχαν. Κύριε Πρόεδρε, Herr President, όπως θα πρέπει να, συζητήσω, να συνηθίσω να σας λέω. Καταρχάς να σας συγχαρώ εξ ονόματος της ομάδας μου για την εκλογή σας ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ευχαριστώ και τον Γέρζι Μπούζεκ για όσα έκανε τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Μπόρεσα να συνεργαστεί μαζί του τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ήταν ιδιαίτερα ικανός και άξιος πρόεδρος και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για σας να ακολουθήσετε τα βήματά του. Κύριε Σούλς, ε, ε, μιλήσατε στο περιοδικό Spiegel και είπατε ότι ε, ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει αποφάσεις, αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Συμφωνώ βέβαια με την άποψή σας, αλλά με κάποια ηρωνία δεδομένου του τρόπου με τον οποίο εκλεγήκατε. Είχατε μια πολύ καλή πλειοψηφία σήμερα το πρωί αλλά δεν ήταν ε, αξιοσημείωτη και θρίαμβος η πλειοψηφία σας, όπως θα παρατηρήσατε, και να ευχαριστήσω και την Ταϊάννα Γόλη και τον συνάδελφο Νίρς Δίβα, που το έκαναν αυτό εκλογές και όχι στέψη. Θα πρέπει ε, να είμαστε περήφανοι, διότι έκαναν προσπάθεια να γίνει πλήρη συζήτηση για την Προεδρία, για το τι ακριβώς ε, εμπεριέχει και τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει. Ο έκανε μια εκλογική εκστρατεία με πολύ χαμηλό προφίλ ως συνήθως και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την εκστρατεία του. Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία για το επόμενο διάστημα στην Προεδρία σας. Η ομάδα μου θα τιμήσει ε, την Προεδρία σα και θα συνεργαστούμε επικοδομητικά μαζί σα παρά τις προφανείς πολιτικέ μας διαφορές. Ε, δεν συμφωνώ με όλε τι δηλώσει που κάνετε σήμερα το πρωί, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε μια άλλη φορά, είμαι βέβαιο, διότι αυτή είναι η φύση τη δημοκρατία. ο καθένα να σέβεται τι απόψει του άλλου, παρά το γεγονό ότι μπορεί και να ερίζουν οι απόψεις μας. Ε, είμαι βέβαιο ότι θα φερθείτε σε όλου με ισότιμο τρόπο και με το δέοντα σεβασμό για ανεξάρτητα από την πολιτική ομάδα στην οποία ανήκουν. Η πρώτη βασική σας δέσμευση θα είναι η εκπροσώπηση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μερικές εβδομάδες και είμαι βέβαιος ότι όλοι οι επικεφαλείς ε, κρατών και κυβερνήσεων ε, θα χαρούν ιδιαίτερα να ακούσουν τι έχουν να πούθουν, διότι δεν ακούγονται και πολλές απόψεις σοσιαλιστών στο Συμβούλιο, επομένως θα θέλουν να ακούσουν και την άποψή σας για τα θέματα αυτά. Σε αυτή τη συνεδρίαση και σε όλε τι άλλες συνεδριώσει, στις οποίε θα πρέπει να παραστείτε ω πρόεδρο, σα εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλέν. Η συνάδελφο Λιωτάρα έχει τώρα εξ να τη ομάδα τη. Παρακαλώ. Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση να αντικαταστήσει κανείς τον πρόεδρό μας Λοταρπίσκι. Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμότατα για την εκλογή σας. Αμέσως ε, πετύχατε την πλειοψηφία αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους ανθυποψηφίους σας. Πραγματικά έκαναν ό,τι μπορούσαν και ελπίζω στο μέλλον να συμβούν πολύ περισσότερα και να μπορέσουν και άλλα να καταθέσουν υποψηφιότητε. Προσωπικά θεωρώ μεγάλο κρίμα που δεν είστε γυναίκα, αλλά τι να κάνουμε, δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να δείξετε και τη γυναικεία σας πλευρά καμιά φορά. Πολλά μέλη σας ψήφισαν, πάρα πολλά του Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιη, <laughs> είμαι βέβαιη ότι το έπραξαν για να σας ευχαριστήσουν, αλλά υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που θεώρησαν ότι θα του δυσκολεύσουμε για τη ζωή του κυρίου Σούλτς διότι εκλέγεστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, σε πάρα πολύ χαλεπούς καιρούς, καιρούς κρίσης. Και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο στην οικονομική και κοινωνική κρίση που διανύουμε. Είμαστε το μόνο ε, άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο από τους πολίτες οι οποίοι ε, πολίτες αγωνιούν μην χάσουν τις δουλειές τους, μην χάσουν τις συντάξεις τους και ανησυχούν αν ε, μπορεί ακόμα το σύστημα υγείας να σταθεί στα πόδια του να μπορούμε να το πληρώνουμε και αγωνιούν και για το μέλλον των παιδιών τους. Ελπίζω να δώσετε φωνή σε αυτούς ακριβώς πολίτες και σας ζητώ να το πράξετε. Ξέρω ότι σε πολλά θεσμικά όργανα Συχνά γίνεται λόγος για χρήματα και το χρήμα και τα μεγάλα συμφέροντα κυριαρχούν αλλά εμείς είμαστε εδώ για τους πολίτες. Πολλές συμφωνίες γίνονται κρυπτό και παραβίστο, όπου ο πολίτης δεν μπορεί ούτε να δει ε, πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να φροντίσετε εσείς να επέλθει μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και να ακούγονται οι διάφορες απόψεις μικρών και μεγάλων ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι είστε πρόεδρος όλων μας. Εμείς ως Ενωτική Αριστερά θα φροντίσουμε να το θέτουμε υπόψη σας. Ελπίζω να ε, έχετε καλή επιτυχία στο έργο σας και με μεγάλη σοφία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεωτάρ. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτά που λέτε ο, ο κύριος Φερχόφστατ λέτε να μην είναι πρόεδρος χωρίς φίλο, η κυρία Λεωτάρ μου λέτε κρίμα που δεν είστε γυναίκα. Τι να κάνω, θα βάλω τα δυνατά μου να ανταποκριθώ σε αυτά που μου ζητάτε. Ο κύριος Φεράτζ έχει το λόγο εξ της ομάδας του. Well, good morning, Mr. Schultz. President Schultz. Καλημέρα κύριε Σούλτ. Πρόεδρε Σούλτ, ξέρω ότι ρόλος μου είναι να σας συγχαρώ. Αλλά επειδή το αποτέλεσμα ήταν γνωστό εδώ και δυόμιση χρόνια, λόγω των συμφωνιών τελικά δεν έχει και πολύ νόημα. Στην σύγχρονη Ευρώπη, όποιο έχει μια θέση εξουσία, θα έπρεπε να αποφασίζεται η απόδοση τη θέση αυτή με μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία. Είμαι σίγουρο ότι θα συμφωνείτε. Τέλο πάντων, ήταν διασκεδαστικό το σημερινό πρωινό, διότι σκέφτηκα τι είδου πρόεδρο θα είναι ο κύριο Σούλτ. Θα είναι ένα ήρεμο, αξιοπρεπή πρόεδρο ο οποίος θα μπορεί να εκπροσωπεί όλα τα μεγάλα κοινοβούλια ανά τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει τις μεγάλες ε, πολιτικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις λεπτομέρειες σαν ένας ε, φιλόδοξος ε, πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι αυτός που γνωρίζουμε από το 2004 ως αρχηγός των σοσιαλιστών ο οποίος πολύ συχνά γκρινιάζει, είναι θυμωμένο, χάνει την ψυχραιμία του, δεν ανέχεται διαφορετικές απόψεις κάποιος ο οποίος προκαλεί όταν υπάρχουν διαφωνίες ε, διενέξεις και συγκρούσεις ο οποίος βέβαια γνωρίζει τα πολιτικά πράγματα στα δάχτυλά του, αλλά δεν του αρέσει και η ελεύθερη αγορά. Είχα πολλά ερωτηματικά λοιπόν και είναι σαφές ότι θα έχουμε δυόμιση χρόνια πολιτικού φανατισμού από την πλευρά της Προεδρίας, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι μόνο σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, μόνο σε μια δημοκρατία της ε, Αφρικής, μια μπανανία θα ήθελε να έχει έναν τέτοιο πρόεδρο για πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου. Αλλά αυτό μας έλαχε. Μπορεί να εκπροσωπώ τη μικρότερη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Σούλτ, αλλά σα διαβεβαιώ ότι είναι μια ομάδα τη οποία θα ιδεώδη και οι απόψει αυτή τη στιγμή απηχούνται από έναν αυξανόμενο ρυθμό πολιτών σε όλη την Ήπειρο. Είμαι βέβαιο ότι θα συμφωνείτε, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσει. Είναι 50-50 πλέον ε, τα ποσοστά. Εάν ε, για να, αν ερωτήσουμε του πολίτε τι θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό ή κακό στοιχείο για τη ζωή του. Δεν είναι ο στόχο να είμαστε κατά τη Ευρώπη. Δεν είναι αυτό η βασική άποψη τη της, ε, ομάδα μα. Πιστεύουμε στην Ευρώπη των κρατών. Θέλουμε Ευρώπη του εμπορίου, τη συνεργασία που να είναι υπεύθυνη. Δεν θέλουμε όμω μία Ευρώπη η οποία θέλει να είναι μία παγκόσμια υπερδύναμη. Δεν θέλουμε μία Ευρώπη την οποία, την, ε, της οποίας να ηγείται ο κύριο Μπαρόζο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη λεγόμενη κοινοτική μέθοδο. Θα κάνω λοιπόν ό,τι καλύτερο μπορώ για να αντισταθώ πολιτικά στην Προεδρία σα κατά τη διάρκεια των 2,5 ετών που έρχονται. Και ελπίζω ότι θα ακούσετε τι δικέ μα απόψει. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει εξ ε, της ομάδας ο κύριος ε, Μάντλενερ. Ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς για τη συμφωνία εκλογής σας που είχε γίνει πριν από δυόμιση χρόνια και σήμερα υλοποιείται. Εξ ονόματος της ε, ομάδας μου σας συγχαίρω. Δυστυχώς δεν κάναμε προεκλογική εξτρατεία και debate. Ε, ο κύβος είχε ήδη ρηφθεί, ε, είναι γνωστό. Και βγήκατε αμέσως από την κάλπη νικητής. Τι να κάνουμε. Πριν από ένα χρόνο αποκαλέσατε φασίστα ένα συνάδελφό μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν αρμόζει κάτι τέτοιο σε ένα δημοκρατικό βουλευτή. Και ποτέ δεν θελήσατε να πάρετε αποστάσεις από αυτή σας τη δήλωση. Και ούτε αρμόζει σε εσά αυτό, δεν σας τιμά. Το θεωρώ μεγάλο κρίμα και ελπίζω ότι είναι ακόμα καιρός να πάρετε πίσω αυτή τη δήλωση. Διότι, Πρόεδρε, δημοκρατία είναι η δημοκρατία μόνο όταν δέχεται κανείς και την αντίρρηση και όχι να χαρακτηρίζει κάποιον φασίστα επειδή διαφωνεί μαζί του. Είμαστε όλοι δημοκράτες μέχρι το μεδούλι, έχουμε εκλεγεί δημοκρατικά και θα πρέπει να μας σέβεστε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την εμπιστοσύνη στα μάτια των πολιτών. Όλο και περισσότεροι πολίτες ζητούν να επανέλθει η εθνική κυριαρχία. Οι μικρές χώρες μπορεί να είναι ε, σε ευημερία και να συνεργάζονται σε ειρήνη, αλλά αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης. Με τη στρατιωτική σημαία του ΝΑΤΟ ε, ακούμε διάφορα ε, για ε, το, στρατιωτικέ τις στρατιωτικές προσπάθειες, αλλά μας έχει εξασφαλίσει στην Ευρώπη ειρήνη. Η σοσιαλδημοκρατία, κύριε Σούλτσα, έχει ε, πτωχεύσει, έχει χρεοκοπήσει. Θα πρέπει ε, να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε όλη την κατάσταση στην Ευρώπη και ελπίζω, κύριε Σούλτς, να είστε και δικός μας πρόεδρος Σούλτς, να γίνετε πρόεδρος και να αφήσετε το σοσιαλδημοκράτη στην άκρη και να γίνετε πλέον υπερκομματικός για να έχετε μια αξιοπρεπή Προεδρία και να ε, ακούτε όλες τις δημοκρατικές απόψεις που εκπροσωπούνται εδώ. Είμαστε δημοκρατικά εκλεγμένοι βουλευτές. Μπορεί να μην ανήκουμε σε κάποια πολιτική ομάδα, αλλά έχουμε τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπολείπους. Και για το μέλλον, Πρόεδρε, Εμείς πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία και στη δύναμη των κυρίαρχων κρατών και όχι στη σοσιαλδημοκρατία. Σας εύχομαι λοιπόν επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και καλό θα ήταν να ακούτε και τις ε, δικές μας φωνές και θα σταματήσει αυτό το τσίρκο μετακόμισης Στρασβούργο, Βρυξέλλες και Τούμπαλιν. Δούμε τι θα γίνει ε, στην επόμενη σύνοδο κορυφή. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία ε, και ελπίζω να επιτύχει τι νέα σα καθήκοντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Πρόεδρος κ. Μπαρόσο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Μάρτιν Σούλτς, αξιότιμοι κύριε και κύριοι βουλευτέ, Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατές μου ε, τα θερμότατά μου συγχαρητήρια για την επιτυχή εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξελέγει και πρώτη φορά Ευρωβουλευτής το 1994. Έκτοτε εντυπωσίασε στο Κοινοβούλιο με την ισχυρή του προσωπικότητα, τις πολιτικές του ικανότητες και την ακαταπώνητη προσπάθειά του για το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Έχει και πολύ σωστά φιλόδοξα οράματα για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Και όντως θα φροντίσει να ακουστεί πολύ πιο δυνατά από ό,τι στο παρελθόν η φωνή του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ο Μάρτιν Σούλτς μπορεί να στηρίζεται στην υποστήριξη ολόκληρη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όντως σήμερα θα πρέπει να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Εκείνοι οι οποίοι σε εθνικό επίπεδο ισχυρίζονται πως η δημοκρατία μπορεί να είναι μόνο εθνική, δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχουμε περάσει ήδη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στον 21ο αιώνα ζούμε. Όσοι αντιστέκονται στην ιδέα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, και της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μάλιστα, επικαλούμενη την εθνική κυριαρχία, παραδίδουν την πραγματική τους κυριαρχία σε κάποιους ανώνυμους παράγοντες των αγορών που δεν υπάγονται σε κανέναν δημοκρατικό έλεγχο. Και όντως, στην περίοδο αυτή κρίσεως, όταν οι μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι όλο και μεγαλύτερες, είναι πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό πλέον, να αγωνιστούμε από κοινού για μια ισχυρή Ευρώπη όλες οι πολιτικές δυνάμεις και γι' αυτό θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή σε όλους τους άλλους και στους άλλους υποψηφίους, την κυρία Γόλης και τον κύριο Ντέβα. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω ειλικρινά βέβαια και τον απερχόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Γιάννη Μπουζέκ. Ο πρόεδρος Μπούζεκ προείδρευσε στο Κοινοβούλιο με έναν τρόπο εντυπωσιακό και επιθαρχημένο σε στιγμές ιστορικών δοκιμασιών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως και επίσης μερικές από τις πιο κρίσιμες ε, πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη την ιστορία της. Η στενή και καλή συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων κατά τα τελευταία δυόμιση χρόνια έθεσαν τα θεμέλια για μια ε, υγιή και γεμάτη εμπιστοσύνη, ειδική σχέση συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οδηγώντα μα σε ένα κοινό κεκτημένο. Όμω, πέραν όλων αυτών, ο πρόεδρο Μπούζεκ ήταν ο, πρώτο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Θεσμικού Οργάνου, ο οποίο προέρχεται από ε, τα κράτη τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ε, μετά την πτώση του σιδηρού παραμετάσματο. Η Προεδρία του ε, ουσιαστικά εκφράζει το όνειρο εκατομμυρίων ανθρώπων που έγινε πραγματικότητα Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. για Μπάρντο. Κυρίες και κύριοι, η ευθύνη μας είναι να θέσουμε πλήρως σε ισχύ τις ε, αποφάσει που λήφθησαν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο ενωμένη. Τα μέτρα τη οικονομική σταθερότητα και τη οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αποτελέσουν τι προτεραιότητέ μα για του ερχόμενου μήνε. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη βασιζόμενη μόνο στην πειθαρχία και τι κυρώσει. Θα πρέπει η Ευρώπη να οικοδομηθεί με γνώμονα την σύγκληση, την αλληλεγγύη και την ελπίδα. Για αυτού ακριβώ του λόγου η ανάπτυξη αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν η ελπίδα να υπερισχύσει εναντί του κινησμού και της απογοήτευσης και να επιβεβαιώσουμε εκ νέου την κοινή μας βούληση να συμβιώσουμε. Πρέπει όμως να απαιτήσουμε και θυσίες και θυσίες οι οποίες θα πρέπει να μοιραστούν με τρόπο ισότιμο. Δεν μπορεί πάντοτε η πλέον αδύναμη και οι μεσαίες τάξεις να καταβάλουν το μεγαλύτερο τίμημα του λογαριασμού που προκύπτει από την κρίση. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα, ένα απαραίτητο στοιχείο για να πετύχει η απόκριση που θα δώσουμε στην κρίση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς που ταυτόχρονα είναι και συναρπαστικοί, πρέπει να εκφράσω λοιπόν τις ε, ευχές μου για επιτυχία μπορείτε να υπολογίζετε στην αμέριστη συνεργασία μας ε, και τη διαρκή συνεργασία μας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε η Ευρώπη να βγει από την κρίση πιο ισχυρή και πιο ενωμένη από ποτέ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα λιγότερα καλά σας λόγια και πάλι για αυτά σας ευχαριστώ. Είναι για μένα συγκινητική στιγμή, για πολλούς φίλους μου επίσης. Και μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε ευχαριστίες μου προς όλους σας. Μια προσωπική παρατήρηση. Όπως είπα, θα προσπαθήσω να είμαι πρόεδρος όλων σας, ανεξαρτήτως πολιτικών ομάδων και πεπιθήσεων είναι και καθήκον αλλά και υπόσχεσή μου. Σας ευχαριστώ. Εσάς κύριε Μπαρόζο. Τα θεσμικά μας όργανα είναι αλληλοσυμπληρούμενα και αυτός ο ρόλος όχι απλώς είναι απαραίτητο, αλλά και ζωτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορείτε να υπολογίζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν τι άλλο στη συντριπτική του πλειοψηφία και σε μένα προσωπικά ως μελλοντικό σας σύμμαχο τη μάχη που δίδουμε για να υποστηρίξουμε την κοινοτική μέθοδο. Κυρίες και κύριοι, spoken uh, τα λόγια σας πραγματικά με συγκινούν. και όλα αυτά που είπατε για μένα. Είναι μεγάλη ευθύνη και πάρα πολύ σημαντικό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να είναι πρόεδρος όλων των μελών του Κοινοβουλίου. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι σοσιαλδημοκράτης παραμένω. Αλλά δεν είμαι ο πρόεδρος της Σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, με πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πάλι το καθήκον μου είναι να υπερασπίζω τα συμφέροντα του Κοινοβουλίου. Και παρακαλώ να αντιληφθείτε. Μια πρόσθετη ακόμη παρατήρηση είναι έντονη αυτή τη στιγμή συγκινησιακά για μένα, αλλά όχι μόνο για μένα, γιατί εδώ στην αίθουσα είναι πολλοί από τους φίλους μου και όχι μόνο μέσα στο ημικύκλιο, επάνω στα θεωρία, φίλοι μου, πρώην δάσκαλός μου, από το σχολείο μου, όταν ήμουν 7 χρονών παιδί, έχουν έρθει κοντά μου, έχουν έρθει φίλοι από την ποδοσφαιρική μου ομάδα που δεν ήταν η πιο επιτυχημένη αλλά πάντως η καλύτερη για μένα στη ζωή μου. Φίλοι μου από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρώην Δήμαρχος, της πόλης μου, ο Τρέχον, δήμαρχος, η προκάτοχή μου και διάδοχή μου ως ε, δήμαρχος ε, του, στη θέση του Δημάρχου του Άχεν και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να τους καλωσορίσω από εδώ στα θεωρία μας γιατί είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Στα γαλλικά. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί πρώην πρόεδροι του Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αλλά και για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η παρουσία σας εδώ. Με μεγάλη χαρά σας βλέπω εδώ απέναντί μου και αντιλαμβάνομαι πόσα χρόνια έχουν περάσει που είμαι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα την τιμή να υπηρετήσω υπό τον κάθε ένα εξιμόνο, πλην του Ενρίκε Μπαρόσο. Γιατί... Μπαρόν. Γιατί... Ε, γιατί ήρθα μετά από τη δική του θητεία ως πρόεδρο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την τιμή που μας κάνατε, σε μένα προσωπικά και στο Κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι, κάτι καινούριο που ήθελα επίσης να σας ε, επισημάνω, κάτι πολύ σημαντικό και για την πολιτική μας εικόνα γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε να εργαστούμε για να βελτιώσουμε την πολιτική μας εικόνα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ίσως, γιατί πλήττεται βαθύτατα η πολιτική μας ομάδα, ε, εικόνα την ώρα που ομιλεί το, ε, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ή των, ε, του Συμβουλίου και μπαίνουν συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα συζητώντας και κάνοντας φασαρία. Λοιπόν, αντί για το δυσάρεστο θέαμα του σφυριού που χρησιμοποιεί ο Πρόεδρος, εγώ αποφάσισα να χρησιμοποιήσω κόδωνα για να σας επαναφέρω στην τάξη. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Λίγα λόγια διαδικαστικά ήταν μόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξή σας. Και πριν να συνεχίσουμε αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα ως ε, νέο εκλεγής πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απευθυνθώ και προς εκείνους που ήταν υποψήφοι μαζί μου, τον κύριο Ντέβα, την κυρία Wallis. Θέλω να σας ευχηθώ και κυρίως γιατί ο αγώνας ο εκλογικός αυτός ήταν τόσο ε, ανοιχτός, τόσο σωστός Όταν είδα το πρωί τα λουλούδια, που, το, τα μπαλόνια που ήταν στολισμένα το κοινοβούλιο, θεώρησα ότι θα ήταν κάποια εκστρατεία για την απελευθέρωση της Γιούλια Τιμοσέγκο, γιατί ξέρετε ήταν το σύμβολο του αγώνα της στα μπαλόνια, αλλά ήταν ο εκλογικός αγώνας του κυρίου Ντέβα. Κυρία Γουόλης, θα ήθελα και εσάς να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε συμβάλει και θα συνεχίσετε φαντάζομαι να συμβάλλετε, όπως ελπίζω, στην, ε, στη συζήτηση του Κοινοβούλιο και ότι θα επηρεάσετε και τη δική μου δουλειά από εδώ, τη θέση του Πρόεδρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω απ' όλα για την ισότιμη και δίκαιη και τίμια αντιπαράθεση και προσβλέπω σε μια πολύ καλή συνεργασία από εδώ και μπρος. Αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι.